Mes chers collègues, je vous propose euh, que nous commencions. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέω να αρχίσουμε. Λέω. Σας καλημερίζω όλες και όλους. Συγχαίρω θερμά όλα τα μέλη που είναι παρόντα εδώ, τα νέο εκλεγέντα και τα απλώς εκλεγέντα. Χαίρομαι που βλέπω πολλά γνωστά πρόσωπα αλλά και άγνωστα και καλωσορίζω λοιπόν τα ιδιαίτερα τα νέα μέλη στην Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων και χαίρομαι που όλοι μαζί αρχίζουμε μια νέα θητεία που είμαι βέβαιη ότι θα αποβεί πολύ ενδιαφέρουσα. Επίσης χαίρομαι που ξαναβρίσκω εδώ και τα μέλη της γραμματείας και τα ευχαριστώ εκ των προτέρων για όλη τη δουλειά που θα κάνουμε μαζί. Επίσης ευχαριστώ επίσης εκ των προτέρων τους διερμηνείς χωρίς τους οποίους δεν μπορούμε να δουλέψουμε αποτελεσματικά. Βάσει του άρθρου 14.1 του κανονισμού ως δεύτερη αντιπρόεδρος, πρώην δεύτερη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμικών προεδρεύω εγώ μέχρι να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, μέχρι να παραδώσω τη σκητάλη. Αρχίζει λοιπόν επίσημα εδώ η συνεδρίασή μας που έχει ως μοναδικό στόχο την εκλογή του Προεδρίου της. Δηλαδή πρώτα του Προέδρου και το μετά των Αντιπροέδρων σύμφωνα με το άρθρο 204 του κανονισμού πρώτα θα εκλέξουμε τον πρόεδρο και μετά τους αντιπρόεδρους. Θα σας πω πρώτα τους ε, αναπληρωματικούς που θα έχουν δικαίωμα ψηφοφορίας εδώ. Το ΕΛΚ μας γνωστοποίησε ότι μερικοί αναπληρωματικοί θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία στη θέση των πλήρων μελών που δεν μπορούν να έρθουν. Τρεις είναι αυτοί. Πιλάρ Αγιούσο, Ιβάνα Μάλετιτς, Βιβιάν Ρέντινγκ που θα αντικαταστήσουν τους κυρίους Μιγκουέλ Αρίας Κανέτε, τον Έλμαρ Μπρόκ και τον Σάιρος Βόλσκι. Μήπως κανείς άλλος αναπληρωματικός ε, πρέπει σήμερα να ψηφίσει γιατί ορίστηκε ως αντικαταστάτης κάποιου πλήρους μέλους. Από την ομάδα του, όχι. Ωραία. Πρέπει τώρα να σας ρωτήσω αν έχετε τις κάρτες σας μαζί σας. Για την περίπτωση που θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε αν δεν μερικοί την έχετε ξεχάσει, έχει, έχουμε ακόμη χρόνο να την φέρουμε. Όχι. Δεν θέλει κανείς να δηλώσει ότι ξέχασε την κάρτα του. Όχι. Αρχίζουμε λοιπόν. Καταρχήν να δούμε αν υπάρχει απαρτία. Υπάρχει προφανώς ένα τέταρτο των μελών δηλαδή και τώρα ζητώ τις υποψηφιότητες. Υπάρχει καμία πολιτική ομάδα που θέλει να παρουσιάσει υποψηφιότητα. Ορίστε κύριε Σαφήν μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω όλα τα νέα μέλη. Εξ ονόματος του ΕΛΚ προτείνω την υποψηφιότητα ως Προέδρου της ΑΦΚΟ της κυρίας Ντανούτα Χούμπνερ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Κυρία Ντανούτα Χούμπνερ, αποδέχεστε την υποψηφιότητά σας. Ναι, δέχομαι. Μήπως τότε υπάρχει καμία άλλη υποψηφιότης από πολιτική ομάδα. Όχι. Όχι. Ωραία. Έχουμε την υποψήφια από το ΕΛΚ. Είναι όπως προβλέπετε και πλήρες μέλος και έχει συμπληρώσει τη δήλωση των οικονομικών συμφερόντων. Αυτές, αυτά είναι τα δύο κριτήρια που απαιτούνται για να μπορεί κανείς να είναι υποψήφιος. Μία και μόνη υποψήφια λοιπόν του ΕΛΚ, η κυρία Ντανούτα Χούμπνερ. Λέω, όπως συνηθίζεται όταν είναι μόνο ένας υποψήφιος, να την εκλέξουμε δια βοής. Voilà. Merci beaucoup. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαίρω την κυρία Ντανούτα Χόμπνερ που μόλις εξελέγει διαβοής πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της παραδίδω αμέσως τη θέση. Uh, Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Αμέσως το επόμενο σημείο η εκλογή των αντιπροέδρων. Ίσως ξέρετε ότι έχουμε τέσσερις αντιπροέδρους. Λοιπόν, υποψήφιος για πρώτο αντιπρόεδρο είναι από την ΓΚΟΕ θα προτείνει η Γκουε μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Εξ ονόματος της Γκουε θα ήθελα να προτείνω τη συνάδελφό μας Βαρβάρα Σπινέλη που δεν έχει μόνο ένα πολύ γνωστό όνομα για την Ευρωπαϊκή Ενωπήση αλλά είναι και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με πολλούς αγώνες. Νομίζω θα είναι πολύ καλή αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως για τον πρώτο αντιπρόεδρο υπάρχει καμία άλλη υποψηφιότητα. Δεν βλέπω. Άρα ρωτώ την κυρία Σπινέλη, δέχεται την πρόταση. Δέχεται την υποψηφιότητά της. Ναι, δέχομαι. Και εδώ ένας υποψήφιος, πάλι διαβοής λοιπόν. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Δεύτερος αντιπρόεδρος. Πρόταση των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε και εμεί εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να σα συγχαρούμε για την εκλογή σας και να προτείνουμε υποψήφιο εκ μέρου τη ομάδα μας για τη θέση του Δευτέρου Αντιπροέδρου, τον κύριο Πέτρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλε υποψηφιότητε. για τη θέση του Δεύτερου Αντιπροέδρου. Κύριε Σπινέλη, θα έρθει να με καθίσει εδώ κοντά μας. Ναι, ξέρετε, διέπραξε ένα το λάθος. Θα ναι, έπρεπε, θα να έχω δηλώσει ότι έχουν κάνει τις σχετικές δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων όλοι οι υποψήφοι παράληψης. Παράληψη. Μπορούμε λοιπόν τώρα και για τη θέση του Ευτέρου Αντιπροέδρου να ε, επικυρώσουμε διαβοή στην εκλογή. Πέντρο Σίλβα, Περέιρα. Περάστε. Και προχωρούμε με την εκλογή του τρίτου αντιπρόεδρου εκ μέρου των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, ο κ. Μέσσερ Σμιτ, παρακαλώ. Ναι, εκ μέρου ομάδα μου έχω την τιμή να παρουσιάσω το υποψήφιο τον κύριο Πουγιαστόφσκι, πρώην Υπουργό Ζαζιτόφσκι. Το παρακαλώ λοιπόν να μας πει αν δέχεται την υποψηφιότητα αυτή. Υπάρχει άλλος υποψήφιος. Επομένως άλλος ψήφιος δεν υπάρχει. Διαβοής. Έχουμε θέσει ακόμα για τους αντιπρόεδρους μας. Βεβαίως. Και ο τρίτος αντιπρόεδρος παρακαλείται να έρθει στο Προεδρείο και προχωρώ στον τέταρτο αντιπρόεδρο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλει να υποβάλει τον κύριο Παόλο Ραντζέλ ως υποψήφιο για τη θέση του Τετάρτου Πρόεδρου. Ευχαριστώ. Δέχεστε την υποψηφιότητα, κύριε Ραντζέλ. Ναι. Έτερος υποψήφιος υπάρχει. Άρα και πάλι διαβοής νομίζω ότι μπορούμε για λόγους και ισότιμης μεταχείρισης. Παόλο, αν έχουμε ακόμα μια θέση ελεύθερη. Έλα και εσύ στο Προεδρείο. Πολλά άλλα θέματα δεν έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Στα διάφορα. Έχουμε και την προσοχή μας συνεδρίας που θα είναι και η πρώτα τακτική στις 22 του μηνός το απόγευμα. Θέλω επίσης να σημάνω ότι έχουμε προβλήματα γιατί υπάρχει σύμπτωση στον προγραμματισμό με άλλες ε, συνεδριάσεις, αλλά θα μας βοηθήσει ο γραμματέα μας, μας να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Και επίσης οι συντηρητικοί μεταρρυθμιστές μας έχουν ζητήσει για ένα λεπτό να τους ακούσουμε χωρίς συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα που αφορά την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι πεπισμένος ότι Η ψηφοφορία αυτή που θεωρείται άλλωστε και μεγάλο επίτευγμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι δημόσια και ονομαστική. Ένα τέτοιο εγχείρημα, ένα διάβημα μάλλον σε σχέση με την τροποποίηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου θα υποβληθεί από πλευρά μα. Αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει προεργασία πριν από το Στρασβούργο γιατί προβλέπετε ότι θα γίνει η, εκλογή, την, ε, ψηφοφορία για την εκλογή του Πρόεδρου της Επιτροπής ε, στην προσεχή σύνοδο. Καλώς λέει η Πρόεδρος, δεν ε, θα γίνει συζήτηση, απλώς όπως σας είπαμε δίνουμε το λόγο για ένα λεπτό στον εκπρόσωπο των στερετικών μεταρρυθμιστών και τώρα κυρίσω το πέρα στην σας, γιατί θα ξανασυναντηθούμε στις 22-3 το απόγευμα, εν τω μεταξύ θα γίνει στη συνεδρία των συντονιστών βεβαίως, αλλά θα ενημερωθείτε.